Αυτό που απαιτείται είναι κοινοτική αλληλεγγύη και συντονισμός δράσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Now, Mr. Madlener. Ο κύριος Μάντλενερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωζώνη